να μην αποφασίζεται στη διάσκεψη των Προέδρων, αλλά συνολικά από όλους τους βουλευτές. Colleagues, I am informed that there was an Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, με ενημερώνουν ότι έγινε πολύ εκτενή συζήτηση και σε μεγάλο βάθο σήμερα το πρωί στη διάσκεψη των Προέδρων και νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το όργανο του Κοινοβουλίου να επιλύει το θέμα και στο μέλλον. Τα σχόλιά σα πάντω έχουν ε, σημειωθεί και ε, προβληματίζουν και άλλου. Αλλά α προχωρήσουμε τώρα, σα παρακαλώ, στι ψηφοφορίε. Κύριε Ράνστορφ, για το ίδιο θέμα είναι. Εάν ναι, ε, όχι, θα περάσουμε στη ψηφοφορία. Κύριε Ράνστορφ, για το ίδιο θέμα θέλετε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Για το ίδιο θέμα. Γνωρίζω ότι το γραφείο Ζαχάρη